Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, διότι έχουμε και τη συζήτηση στην Ολομέλεια και ορισμένοι συνάδελφοι πρέπει να αποχωρήσουν, γιατί προβλέπετε να μιλήσουν στην Ολομέλεια. Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους. Μεταδίδεται μέσω διαδικτύου η σημερινή μας συνεδρίαση. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση ημερήσιας διάταξης. Σε ποιο από τα δύο μικρόφωνα μιλήσω, το δεξί ή το αριστερό. Το αριστερό. Πρώτο λοιπόν σημείο της ημερήσιας διάταξης, η έγκρισή της σας έχει διανεμηθεί ήδη από τις 30 Ιουνίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, δεν έχουμε λάβει καμία αντίρρηση μέχρι στιγμής και κανένα αίτημα τροποποίησης, επομένως εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσεις τη Προέδρου. Όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση των συντονιστών, πέρα από τη σημερινή συνεδρίαση σήμερα θα έχουμε και μια συνεδρίαση στις 15 Ιουλίου μισή μόνο μέρα. Έχουμε λοιπόν μια συνεδρίαση μόνο το πρωί στις 15 Ιουλίου. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να έρθετε στη συνεδρίαση αυτή γιατί θα έχουμε τον Υπουργό Νίκολα Σμίτ ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου και επίση θα έχουμε μαζί μα και τον πρόεδρο τη Επιτροπή των Περιφερειών, ο οποίο θα συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρία στις 15 Ιουλίου. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξη, ανακοινώσει τη Πρόεδρου σχετικά με τι συστάσει των συντονιστών. Στην τελευταία λοιπόν συνεδρία των συντονιστών καταλήξαμε σε κάποιε συστάσει οι οποίε πρέπει να εγκρίνουμε σήμερα. Σα έχουμε διανύμει επίσης τα ονόματα των στακτών γνωμοδοτήσεων, γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΑΦΕ, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των Εθνών, πώς μπορούμε να πετύχουμε καλύτερους στόχους όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Ο κύριος Ντέβιτ Μακάλιστερ από το ΕΛΚ θα είναι ο στάκτη γνωμοδότησης. Γνωμοδότηση επίσης να αφορά την ετήσια έκθεση 2014 για την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση της απάτης. Ο στάκτη γνωμοδότησης θα είναι από τους συνταλιστές, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τις δύο αυτές συστάσεις των συντονιστών. Έχουμε λάβει επίσης και δύο προτάσεις ψηφισμάτων τις οποίες τις συζητήσαμε και αυτές στις συνεδρίες των στονιστών, έχουμε μια πρόταση ψηφίσματος για την εγκατάλειψη της στρατηγικής καλύτερης νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την πρόταση αυτή ψηφίσματος παρουσίασαν η Σοφή Μοντέλ και ο Ντομινίκ Μπίλντ. Η πρόταση των συντονιστών είναι να μην δοθεί αυτόνομη συνέχεια στην πρόταση αυτή. Ενδεχομένως αν επιμείνουν οι δύο αυτοί συνάδελφοι θα μπορούσαμε να εντάξουμε την πρόταση αυτή στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη νέα διαθεσμική διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία και έχουμε και μια δεύτερη πρόταση ψηφίσματος για την ε, επανεγκαθίδρυση της δημοκρατίας στην Ευρώπη πρόταση ψηφίσματος που έχει υποβάλει η κυρία Μαριλεπέν, ο Φλωριάν Φιλιππό, ο Ντομινίκ Μπίλτ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Όσον αφορά αυτή την πρόταση ψηφίσματος ε, εγκρίθηκε η ίδια απόφαση με του, από τους τονιστές να μην δοθεί αυτή τη στιγμή κάποια συνέχεια. Θα μπορούσε ενδεχομένω και αυτή η πρόταση ψηφίσματος να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της συζήτησης που γίνεται για την έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Γκί Φερχόφστατ. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν και γι' αυτό αντιρρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνονται οι συστάσεις των συντονιστών. Να σας πληροφορήσω επίσης ότι έχει γίνει μία αλλαγή, μάλλον Έχουμε μια συνεδρίαση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προβλέπεται για την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 2 και 4 στις 3 και 4 το μεσημέρι και θα λάβει χώρα στο κτίριο του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Θα συναντηθούμε λοιπόν στις 2 η ώρα το μεσημέρι στην κεντρική είσοδο του α, Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρέπει να σας πω ότι οι συντονιστές έχουν υποβάλει ένα πολύ μακρύ κατάλογο συμμετεχόντων. Πρέπει να σας πω ότι η συνεδρίαση θα γίνει μόνο στα αγγλικά ενδεχομένως θα μπορούσαν ε, οι συντονιστές να υποβάλουν και ένα κατάλογο ομιλητών με μια συγκεκριμένη σειρά μετά από προτάσεις των ίδιων των πολιτικών ομάδων. Δεν ξέρω λοιπόν αν οι ίδιοι συντονιστές θα μπορούσαν να επιληφθούν λίγο του ζητήματος αυτού. Ποιος θα συμμετέχει και ποιος θα πάρει το λόγο και ποιος θα μιλήσει με ποια σειρά. Αυτό λοιπόν αποφασίσαμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία μας. Ένα έγγραφο πρόκειται να ψηφίσουμε. Γενικός Προπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2016. Μας απασχόλησε η έκθεση αυτή όλο τον προηγούμενο μήνα και το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι υποβάλλατε πολλές τροπολογίες, ότι εξετάσαμε τις τροπολογίες αυτές, είχαν να κάνουν κυρίως με τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία πρότειναν οι πράσινοι. Έχουμε και κάποιες τροπολογίες από την συγγήτρια και τροπολογίες από άλλα μέλη της ΑΦΚΟ και έχουμε και μια προφορική τροπολογία. Δεν υποβλήθησαν πάντως τροπολογίες όσον αφορά την ίδια την γνωμοδότηση της ηγήτριας. Σας έχει δοθεί λοιπόν ο κατάλογος ψηφοφορίας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Θα ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. 18 ψηφίσαντες. Θα σας προσθέσουμε εφόσον χρειαστεί. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία, τροπολογία 7 υπέρ παρακαλώ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση και τροπολογία 7. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 2 υπέρ και 17 κατά. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Ναι, δεν καταλάβετε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι με τροπολογία 3. Λοιπόν, τροπολογία 3 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 17 υπέρ, 2 κατά, 18 υπέρ μάλλον και 2 κατά. Σας ευχαριστώ πολύ, εγκρίνεται. Σας υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε ακόμα αυτή την προκαταρκτική εξέταση για τα πιλωτικά προγράμματα, η οποία πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανεξάρτητα δηλαδή από την έκβαση της ψηφοφορίας αυτής, αν το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρνητικό, δεν θα δοθεί συνέχεια στα πιλωτικά προγράμματα. Πάντως εσείς ατομικά ή ως πολιτική ομάδα μπορείτε να υποβάλλετε εκ νέου τις σχετικές τροπολογίες. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης, η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε εδώ πέρα έχουμε δύο εισηγητές, είναι ο Γιώ Λάινεν από τους συνταλιστές και δημοκράτες και υποφαινόμενοι για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα μπορούσα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση και συνέχεια θα δώσω το λόγο στον Γιώ. Θα μπορούσα να πω λοιπόν ε, λίγα πράγματα για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ο εκλογικός νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις και για ποιο λόγο θεωρούμε ότι αυτός ο εκλογικός νόμος είναι πολύ σημαντικός. Θα συμφωνείτε φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και ιδίω μετά την έναρξη της α, συνθήκης της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύξησε τις αρμοδιότητές του στην έγκριση αποφάσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδυναμώθηκε λοιπόν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεωρήσαμε ορισμένοι ότι κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του συστήματος έγκρισης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ως παρόχος δημοκρατικής νομιμοποίησης στα πλαίσια του συστήματος λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει πραγματικά να μπορεί να αποκριθεί στις νέες του αυτές αρμοδιότητες και στο υψηλό επίπεδο ευθύνη. Και γι' αυτό λοιπόν προκειμένου να κάνουμε πραγματικά υπόλογο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βελτιώσουμε και τον εκλογικό νόμο. Θα πρέπει δηλαδή μέσω του εκλογικού νόμου να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε λίγο τη διασύνδεση ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι συμμετέχουν σε μια εκλογική διαδικασία και οι οποίοι εκλέγουν δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους. Διασύνδεση λοιπόν ανάμεσα σε αυτό το γεγονός και το θεματολόγιο το οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στον εκλογικό νόμο και για λόγου δημοκρατικής νομιμοποίηση και λογοδοσία. Ξέρω ότι έχουν γίνει πάρα πολλέ αλλαγέ μέσω των διαφόρων συνθήκων όσον αφορά την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όσον αφορά τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δυστυχώς δεν είχαν γίνει απαραίτητες ε, προσαρμογές όσον αφορά τον εκλογικό νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτή τη στιγμή εκλογικά συστήματα τα οποία είναι συνονθήλευμα τελικά πολλών διαφορετικών εθνικών διατάξεων όσον αφορά την εκλογική διαδικασία. Έχουμε πολλούς λοιπόν εθνικούς κανόνες οι οποίοι ε, πραγματικά κυριαρχούν στην όλη διαδικασία η οποία θα έπρεπε να είναι περισσότερο ευρωπαϊκή. Η δική μου άποψη λοιπόν είναι και ελπίζω ότι συμφωνεί και ο είναι Λάινεν ότι θα πρέπει να καταστήσουμε την όλη διαδικασία πιο ομοιόμορφη, να έχουμε περισσότερες κοινέ αρχές στην ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία, να καταφέρουμε να επιφέρουμε λοιπόν τις απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε μία πιο ορατή, προβεβλημένη βάση όσον αφορά τη δημοκρατική αυτή διαδικασία που καταλήγει τελικά στην ανάληψη πολιτικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την άποψή μου λοιπόν ο εκλογικό νόμος δεν είναι μια τυπική απλώς διαδικασία αλλά στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενώπιον των νέων προκλήσεων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της μεγαλύτερης ανάγκη για δημοκρατική νομιμοποίηση ο εκλογικός νόμος και το γυκλό σύστημα διαδραματίζει ένα ουσιαστικό ρόλο. Και οι προσπάθειες λοιπόν που καταβάλαμε με το Γιώ Λάινεν ήταν ακριβώς αυτό, να καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε αυτούς τους α, συνεκτικούς δεσμούς που απουσίαζαν και θα πρέπει το εκλογικό νέο σύστημα αυτό να αποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο Αναφερόμαστε στην αρχή της έκθεσης σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ήδη τα έχουμε συζητήσει με εσά και περιοριζόμαστε προς το τέλος της έκθεσης σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, σε κάποια ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικά και πιο ουσιώδη όσον αφορά τις βασικές αυτές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τον Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο. Του τον να σου δώσω τώρα σε εσένα το λόγο, Γιώ. Ευχαριστώ Δανώτα Ότο κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την καλή συνεργασία των τελευταίων εβδομάδων για το θέμα αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει Brexit ή Brexit. Αλλά εκλογές, ευρωεκλογές θα γίνουν οπωσδήποτε και το αργότερο το 2019. Υπάρχει λοιπόν ευρύτατη συνένεση ότι οι όροι αυτών των προσεχών ευρωεκλογών θα πρέπει να βελτιωθούν είπε και η Πρόεδρος ότι από το 1976 και, το σχετικό, και τη σχετική πράξη για τις εκλογές του 1976 δεν έχει υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Εμεί θέλουμε να είναι πιο ορατές οι εκλογικές αναμετρήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να είναι πιο ε, σαφής η συμμετοχή των κομμάτων και πιο ελκυστική η συμμετοχή των πολιτών. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία λοιπόν που έχουμε προτείνει με, ένα, ε, με μια διαδικασία σε δύο βήματα οι δύο στάδια, καταρχάς με την πρόταση για την τροποποίηση της ε, πράξης της σχετικής με τις εκλογές σε πρώτη φάση και ίσως σε μεταγενέστερη φάση ενδεχομένως και με αναθεώρηση των συνθήκων ή πάντως με, μια ευρύτερη, με έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο βήμα. Πολύ σύντομα λοιπόν, μια και το έχουμε ξανασυζητήσει, θεωρούμε πως τα εθνικά πολιτικά κόμματα που ανήκουν σε μια ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια πρέπει να γίνονται ορατά και στο ψηφοδέλτιο να μπορεί δηλαδή ο πολίτης πάνω στο ψηφοδέλτιο να αναγνωρίζει την ε, υπαγωγή του εθνικού του κόμματος σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Να γίνει αυτό πιο ορατό και ενδεχομένως και στο ε, εκλογικό υλικό, στο, στα φυλάδια της, τα ενημερωτικά και διαφημιστικά, να είναι και αυτό πιο ορατό. Να είναι πιο ορατή δηλαδή η ευρωπαϊκή διαδικασία. Επίσης η σοβαρότητα της ε, προβολής των υποψηφίων. Προτείνουμε λοιπόν προθεσμία για την κατάθεση των εθνικών εκλογικών ε, των καταλόγων υποψηφίων της λίστας της εκλογικής να είναι 12 εβδομάδες πριν από τις εκλογές για τελευταία στιγμή δεν είναι σοβαρό να κατατεθένται τα ονόματα των υποψηφίων. Ε, προτείνουμε επίσης τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να προτείνουν και αυτά τους ε, προβεβλημένους υποψηφίους 12 εβδομάδες πριν. Ξέρουμε ότι δεν το πράττουν όλα τα κόμματα, ότι δεν υποβάλλουν δηλαδή υποψηφίους ε, για τη θέση του προβεβλημένου υποψηφίου, του candidate, αλλά πάντως ε, αυτά που καταθέτουν τέτοιες υποψηφιότητες θα πρέπει να τις καταθέτουν 12 εβδομάδες τουλάχιστον πριν από τις εκλογές. Και επίσης στην εποχή του διαδικτύου και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον θα υπάρχει ασφαλώς όλο και περισσότερη διαδικτυακή ψηφοφορία και ψήφους και άρα θα θέλαμε να προτείνουμε στα κράτη, στο βαθμό που διασφαλίζεται το απόρριτο της ψήφου και μια πρόσκοπτη διαδικασία εκλογής και τη χρήση του διαδικτύου ως προοπτική. Αν, ε, διαπιστώνουμε επίσης ότι δεν επιτρέπεται η επιστολική ψήφος σε όλα τα κράτη, αλλά στα περισσότερα ναι. Προτείνουμε λοιπόν να ε, εξασφαλιστεί η επιστολική ψήφο σε όλα τα κράτη. Επίσης δεν υπάρχει για όλα τα κράτη δυνατότητα της ψηφοφορίας των πολιτών που κατοικούν στο εξωτερικό ε, μέσω των προξενικών αρχών ή καταστημάτων. Προτείνουμε λοιπόν και αυτό να καταστεί δυνατό. Από Πέμπτη έως Κυριακή γίνονται οι εκλογές. Για τις εκλογές επίσης και την Κυριακή υπάρχουν διαφορετικές ώρες που ε, σταματάει η ψηφοφορία, που κλείνουν οι κάλπες. Είναι αυτό ένα πρόβλημα φυσικά γιατί μπορεί σε μια χώρα να έχουν κλείσει οι κάλπες και να αρχίσουν να κοινώνονται αποτελέσματα και γι' αυτό προτείνουμε ώρα 9 κεντρικής Ευρώπης, 9 το βράδυ, συμβιβαστικά, να οριστεί λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τις διαφορετικές ε, ε, ατράκτους ε, τις χρονικές που έχουμε στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, κεντρικά, ανατολικά ή δυτικά. αλλά πάντως 9 το βράδυ, 21 η ώρα κεντρικής Ευρώπης να τελειώνει την Κυριακή ψηφοφορία. Θέλουμε επίσης να έχουμε έναν τρόπο αξιολόγησης και συγκρισιμότητας της εκλογικής πράξης και των εκλογικών ε, πιθανοτήτων της πιθανολόγησης της εκλογιμότητας στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν στα περισσότερα κράτη όρια ε, εκλογικά για την είσοδο στη Βουλή που είναι το 3% επιτοπλίστων, σε κάποια είναι ανάμεσα στο 3% και στο 5%. Υπάρχουν επίσης η Ισπανία και η Γερμανία που έχουν διαφορετικά ε, συστήματα και μπορεί να χρειαστεί και ο, με, τον, με, τον, με την εισαγωγή αυτού του ελάχιστου ορίου και η, ο υπολογισμός του ορίου αυτού όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό, υποπεριφερειακό, καλύτερα επίπεδο. Στη Γερμανία υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει και στην Ισπανία λόγω της περιφερειακής δομής. Με αυτά τα στοιχεία λοιπόν οι προτάσεις μας και όπως είπε και η Πρόεδρος θα έχουμε περισσότερη ορατότητα, σοβαρότητα και ενδεχομένως συμμετοχή στις ευρωεκλογές των πολιτών. Ταυτόχρονα προσεγγίσουμε περισσότερο τους όρους της ισότητας για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ε, Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σέπφλιν. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο για μια πολύ χρήσιμη, πολύ πλήρη έκθεση. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, θέματα τα οποία συζητάμε εδώ και χρόνια, αλλά θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις Πιστεύω πως αυτή η ελάχιστη προθεσμία των 12 ε, εβδομάδων είναι καλή ιδέα. Τώρα το αν θα είναι 12, 16, 14 δεν έχει καμία σημασία αρκεί να ακολουθούμε όλη την ίδια τακτική. Νομίζω αυτό είναι το πιο δίκαιο. 12 εβδομάδες για μένα είναι εντάξει. Και πρέπει να σας πω πως το υποχρεωτικό κατόφλι κάποιου ποσοστού για την είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λειτουργήσει πολύ καλά σε εθνικό επίπεδο. Θα μπορούσε λοιπόν και πανευρωπαϊκά να λειτουργήσει. Για τις υποψηφιότητες αυτές οι 12 εβδομάδες νομίζω κάνουν την όλη διαδικασία πιο δίκαιη παρόλο που ενδεχομένως κάποιοι ήδη θα υποστηρίξουν μια υποψηφιότητα πολύ πριν τις 12 εβδομάδες ε, έτσι ώστε να μπορούν την υποψηφιότητα αυτή να την υποστηρίξουν και να την προωθήσουν Εν το 12 είναι εντάξει. Στην παράγραφο 7 ε, για όσους κατοικούν σε τρίτη χώρα και είναι πολίτες ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής κτλ. Τι ακριβώς τους απαγορεύει από το να το κάνουν σήμερα. Γιατί η εμπειρία που έχω από την Ουγγαρία, εάν κάποιος θέλει να πάει στο προξενείο του, ε, μπορεί να ψηφίσει ας πούμε στο ουγγρικό προξενείο εκεί που βρίσκεται. Υπάρχουν κάποια μέρη στον κόσμο στα οποία δεν υπάρχει προξενική εκπροσώπηση, αλλά νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δώσουμε ε, κάποιο χρόνο στο κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω, να συμμετέχουμε μάλλον μέσω ίντερνετ ε, στις εκλογές. Υπάρχει βέβαια το, πρόβλημα των χρονικών ε, προθεσμιών για το πόσο θα μπορεί, κατά πόσο θα μπορεί κανείς να ψηφίσει μέσω ίντερνετ και αν ε, αυτό γίνεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αν οι ψηφοφορίε που γίνονται σε τρίτες χώρες θα γίνονται νωρίτερα, πώς θα γίνεται η καταμέτρηση. Είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τα τελικά αποτελέσματα. Στην πέμπτη παράγραφο που λέει πως θα πρέπει μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, να έχουν ε, λήξει ψηφοφορίες ε, ε, σε όλες τις χώρες πρέπει να σας πω πως όλοι ξεκινούν σε διαφορετική χρονική στιγμή και θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, δηλαδή θα πρέπει να είναι 9 με 9, θα πρέπει να είναι 12 ώρες ανεξάρτητα από το τι ώρα κλείνει. Είναι μία λεπτομέρεια την οποία θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και ίσως ε, καλό θα ήταν να υποβάλουμε και κάποια συγκεκριμένη τροπολογία. Για την ελάχιστη ηλικία των 16 ετών δεν έχω πρόβλημα να πω όμως το εξής. Κοιτάξτε, οι πάνω από τα 65 ή 70 ε, είναι όλο και περισσότερες χώρες μας και δυσκολεύονται πάρα πολύ να προσεγγίσουν τα εκλογικά κέντρα. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε για την ψηφοφορία μέσω ίντερνετ είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω για το κατά πόσο οι πάνω από τα 75-85 έχουν πρόσβαση και ξέρουν πώς να ε, ψηφίζουν μέσω ίντερνετ. Νομίζω ότι ε, γι' αυτό πρέπει κανείς να είναι αρκετά εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Ίσως κάποιες ειδικέ διατάξεις έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν τα άτομα αυτά σε εκλογικό κέντρο αν είναι μεγάλες ηλικίε, αν πραγματικά είναι αποφασισμένοι να ψηφίσουν και να το προσθέσουμε και αυτό στις διατάξεις μας. Νομίζω πάντως πως η έκθεση είναι πολύ χρήσιμη και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Μερσέδες είναι η επόμενη μιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Και εγώ εν γέννη συμφωνώ με τις επιλογές που κάνατε στην έκθεση αυτή και γενικότερα η ιδέα αυτή που προβάλλεται το ότι θα πρέπει δηλαδή να καταφέρουμε να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά τον υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο. Ένα σημείο πάντως το οποίο προκαλεί κάποιες αμφιβολίες δεν νομίζω ότι στον υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο υπάρχουν δεσμευτικές διατάξεις όσον αφορά τα όσα λέγονται στο κείμενο εδώ πέρα για το φύλλο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν κάποιους μπλοκαρισμένους, μπορούμε να πούμε, εκλογικούς ε, καταλόγους. Και επομένως ε, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποφασίσουν σε καθαρά εθνικό επίπεδο αν ε, η συμμετοχή θα είναι με περισσότερους άνδρες ή περισσότερες γυναίκες. Όταν έχουμε όμως ένα σύστημα με προτιμησιακή ψήφο νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή των φύλων όσον αφορά την σειρά που ακολουθείται στον κατάλογο αυτό. Δεν ξέρω τι υφίσταται στα πλαίσια του εκλογικού νόμου, ενδεχομένω να κάνω λάγο, λάθος, ενδεχομένω εσείς όμως να επιλέξατε να μην ασχοληθείτε συνειδητά με το ζήτημα αυτό, που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γιατί νομίζω ότι σε κάθε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε αυτή την καλύτερη ισορροπία των δύο φύλων και να μην εναπόκειται αυτό μόνο στην εθνική νομοθεσία. Εγώ για παράδειγμα θα υποβάλω μία τροπολογία μαζί με τον συνάδελφο Σέπφλιν. Νομίζω ιδίω ότι για το ζήτημα αυτό θα πρέπει εν μη άλλο να γίνεται μία μνήα στην ε, έκθεση. Να λέμε δηλαδή ότι ανάμεσα στους στόχους που θέλουμε να προωθήσουμε θα υπάρχει και αυτός. Ευχαριστώ, Χέρμουντ Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά και και τον Γιώ Λάινεν για την υποβολή της πρότασης. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά κατ' ουσίαν. Πριν όμως ε, επικεντρωθούμε σε ορισμένε πτυχές, θα ήθελα να κοιτάξουμε τι ακριβώς είναι η κατάσταση μέσα στην οποία κοιτάμε την αναθεώρηση του εκλογικού δικαίου. Μίλησε λοιπόν για δύο βήματα ο Λάινεν. Μία πρώτη φάση για κάποιες μικρές αλλαγές χωρίς τροποποίηση και μετά περισσότερο χρονικό διάστημα με πιο μακροπρόθεσμες αλλαγές που θα σήμαιναν και αναθεώρηση συνθήκης. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε όμως περισσότερη παρουσία εμείς ως, παρησία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι υπόθηκε και στην αρχή των παρεμβάσεων ότι επαπειλείται Brexit ή και Brexit οι τραγικές, ε, τρα, δραματικές μάλλον στιγμέ στην Κροατία ή πολλά πολύ σοβαρά προβλήματα στην Γιατί λοιπόν να πάει να ψηφίσει ο πολίτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν δεν αναγνωρίζεται περισσότερο ότι μετράνε τα συμφέροντα του πολίτη στην πλάστικα των αποφάσεων της ευρωπαϊκή Ένωσης. Εμείς λοιπόν είμαστε ως δομή το άμεσα εκλεγμένο όργανο αυτό δηλαδή το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει τις προσδοκίες του ψηφοφόρου για να ξανακερδίσει αυτόν τον ενθουσιασμό για τη δημοκρατία, τη συμμετοχή, την υποστήριξη και τις προκλήσεις που σημαίνει, σημαίνει η συμμετοχή των πολιτών στο δημοκρατικό γίγνεσθε. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή Ξέρω πολύ καλά, καλύτερα από όλου, ότι πολύ λίγοι θέλουν να αγγίξουν θέματα αναθεώρηση συνθήκων, αλλά πάντω, έστω μέσα σε κάποιε αιτιολογικέ σκέψει, θα πρέπει να δηλώσουμε ότι εμεί δεν θέλουμε να παραβλαφθεί το ευρωπαϊκό μέλλον και το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά ότι θέλουμε παρόλα αυτά να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αυτές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για το εκλογικό δίκαιο. Δεύτερον, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν αλλάζει με τις νέες προτάσεις τίποτα ως προς το γεγονός ότι οι εκλογές γίνονται σε εθνικό επίπεδο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι εθνικές εκλογές για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το σημείο νομίζω πρέπει να το καταδείξουμε πάνω απ' όλα και να δώσουμε και τα δικά μας ορόσημα, να τοποθετηθούμε σε σχέση με αυτό και άρα να συνδέσουμε τα σημεία 1 και 3 για μια δυνατότητα, για ένα ενδεχόμενο διαφορετικής οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας. Και έτσι θα συμφωνήσω με εκείνους που μπορεί να λένε ότι ναι, το 7 είναι ίσως ε, ορθό και πρέπει να το επιδιώξουμε, όσο δύσκολο και μπορεί να φαίνεται αλλά νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η απλούστερη απεικόνηση της εκλογικής διαδικασίας για να αντιλαμβάνεται και ο πολίτης ότι ψηφίζει ευρωπαϊκά και όχι εθνικά. Γι' αυτό και το θέμα της ηλικία, γι' αυτό και το θέμα της ε, ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να το απαιτήσουμε, αλλά ή μη τι άλλο να υπάρξει μια αναγνώριση και με βάση τα εφιστάμενα εκλογικά συστήματα και τους νόμους που ισχύουν στα κράτη-μέλη ε, μπορούμε να βρούμε μια λύση που να επιτρέπει περισσότερη εξισορρόπηση της εκπροσώπησης των φύλων. Αυτό θα ήταν μια λύση προς την ορθή κατεύθυνση. Και κλείνοντας, μια σκέψη που είναι περισσότερο ερώτηση για το σημείο 1 συγκεκριμένα εκεί που λέγεται ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την έννοια της ηθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα πρέπει να στραφούμε στο ζήτημα διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ε, θα ερωτήσω, έχουμε υπόψη το better regulation, την καλύτερη διακυβέρνηση ή μάλλον καλύτερα τις καλύτερες νομοθετικές ρυθμίσεις, έχουμε την καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση, αυτά τα πράγματα τα έχουμε υπόψη σημαντικά, δηλαδή νομοθετήματα τα οποία έχουν οπωσδήποτε συσχετισμό και με την εκλογική διαδικασία. Σε όλα αυτά θα καταθέσω τις τροπολογίες μου. Σας ευχαριστώ. Helmut, ε, very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χέλμουτ. Ε, Επόμενος ο μιλητής ο κ. Χαουρέγγι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συνταχθώ με τις ε, ευχαριστίες όσων μίλησαν ε, πριν από μένα για τον τρόπο που και ο κύριος ε, Τζολάινεν και η πρόεδρος αντιμετώπισαν το θέμα αυτό. Έχω μία μικρή παρατήρηση να κάνω για το δημοκρατικό σύστημα και μία παράσταση και για μία παρατήρηση που έγινε λίγο στα παρεπόμενα ε, λόγω των πρόσφατων εξέλιξεων θα πρέπει στη δημοκρατία να συμπεριλάβουμε και την εξής παρατήρηση. Τα όσα μας επηρεάζουν όλους δεν πρέπει να αποφασίζονται από δημοψηφίσματα ενός. Μιλάμε για πολιτική εντολή και όταν μιλάμε για προβλήματα που επηρεάζουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να επιλύονται όσο δημοκρατικό και αν μας φαίνονται από ένα δημοψήφισμα που γίνεται μόνο σε ένα τμήμα του συνόλου. Το λέω ως κανόνα γιατί εδώ έχουμε κάποιες ε, εθνικές κυριαρχίες που ενδεχομένως θα ε, συγκρούονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μπορεί να έχουμε σήμερα δημοψήφισμα στην Ελλάδα, αύριο δημοψήφισμα στη Γερμανία και να ξεκινήσουν κάποιες συγκρούσεις εθνικής κυριαρχίας όταν θα έπρεπε αυτό να αποφασίσετε περισσότερο από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η μικρή παρατήρηση που θέλω να κάνω στη συζήτηση περί δημοκρατίας και δημοκρατικότητας. Έχω και ένα μεθοδολογικό πρόβλημα με αυτά που παρουσιάζεται κύριε συγητές. Εάν πρόκειται όντως να ακολουθήσουμε μια διετή διαδικασία, δηλαδή ε, να κάνουμε μια ρεαλιστική τροποποίηση του εκλογικού συστήματο σήμερα και παρόλα αυτά αφήσουμε τα πιο οραματικά σχέδια για μια επόμενη ε, μεταρρύθμιση που παραπέμπουμε στις καλέντες των Ρωμαίων, τότε ενδεχομένως χάνουμε μια ευκαιρία, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σόλτς, χάνουμε μια ευκαιρία εμείς να εκφράσουμε μια κοινή θέση για αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε να αποτελεί τον Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο. Δεν πρόκειται για πρόβλημα συνθήκων. Έχει να κάνει με τη βούληση των ε, εθνικών κρατών να τροποποιήσουν τις εθνικές νομοθεσίες για τις ε, εκλογές και να ακολουθήσουν ένα σύστημα ευρωπαϊκό. Θα πρέπει λοιπόν να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο για να μορφώσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία εδώ. Άρα λοιπόν τι θα γίνει, θα παραιτηθούμε από όλους μας τους ε, στόχους. Προσωπικά και εκφράτω στην ομάδα μου να σας πω πως δεν αισθάνομαι άνετα απορρίπτοντας τροπολογίες που υποβάλλουν άλλες ομάδες για θέματα με τα οποία εγώ συμφωνώ. Για παράδειγμα, ε, ισότητα των φύλων, ε, κοινά ψηφοδέλτια. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό συνενετικά γιατί αυτά τα θέματα δεν αφορούν μόνο ένα-δύο κράτη, αποτελούν τους βασικούς κανόνες του δημοκρατικού συστήματος. Εάν πούμε λοιπόν πως η έκθεση αυτή που παρουσιάζουν οι συνάδελφοι θα συμπεριλάβει τροπολογίες τις οποίες εμείς θα απορρίψουμε για παράδειγμα τα ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια ή η κοινή εκλογή κατάλογη ε, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να δούμε με σοβαρότητα για το γεγονός πως συμφωνούμε ή διαφωνούμε δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μία απλή απόρριψη. Να σας παρακαλέσω και κάτι. Θα μπορούσαμε τις προθεσμίες για τις τροπολογίες να μην τις έχουμε για τις 29 Ιουλίου, γιατί είδα το πρόγραμμα και θα ήθελα να μου πείτε αν μπορούμε να παρατείνουμε την προθεσμία για τροπολογίες μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου για τη συγκεκριμένη έκθεση. Uh, η Redding είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες αυτής της ε, έκθεσης για ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο. Μήπως είναι υπερβολικά ρεαλιστικό, μήπως θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει λίγο παρακάτω. Αυτό είναι μία παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς γιατί με κάποιες εξαιρέσεις το κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μας θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τα κράτη-μέλη. Και νομίζω πως αυτό είχαν κατά νου και οι εισηγητές. Συμφωνώ. Συμφωνώ με τις 12 εβδομάδες και συμφωνώ με τα υποχρεωτικά κατόφλια εισόδου, αλλά τι γίνεται με την υποχρεωτική ψηφοφορία. Θέλετε να δούμε πιο οραματικά το μέλλον. Ελάχιστοι ψηφίζουν. Ξέρω ότι σε κάποια κράτη-μέλη είναι υποχρεωτική ε, είναι υποχρεωτικό να ψηφίσει κανείς, κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν είναι. Εάν θέλει λοιπόν κανείς να οραματιστεί, ίσως θα μπορούσαμε να προτείνουμε να είναι υποχρεωτική η προσέλευση στις ευρωεκλογέ. Θα έπρεπε ήδη οι κανόνες να ε, ισχύουν για τους επικεφαλείς ε, των ψηφοδελτίων όπως και για τους απλούς υποψηφίους και θα συμφωνήσω με την πρόταση πως οι επίτροποι που θα ήθελαν να κατέβουν σε εκλογές θα πρέπει να θεωρηθούν ε, ως απληθνητοί και όχι ε, σαν να μεταφέρουν ε, κάποια βαριά ασθένεια, ε, αντιμετώπιση της οποίας έτυχα εγώ όταν κατέβηκα στις εκλογές παρόλο που ήμουν επίτροπος. Τώρα, ε, ψηφοφορία ταχυδρομική, μέσω ίντερνετ, αυτές οι δυνατότητες σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν και επειδή συμφωνώ με τα όσα ήδη υπόθηκαν, πάντα είναι εθνικές οι ψηφοφορίες, ακόμα και αν ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές, είναι πάντα εθνική η ψηφοφορία, οπότε οι καινοτομίες δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά εκτεταμένες γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει να ψηφίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν έχουν συνηθίσει να ψηφίζουν, γιατί νομίζω πως σε κάποια κράτη-μέλη ο κόσμος απλώς αγνοεί το γεγονός πως γίνονται ε, ψηφοφορίες και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις ευρωεκλογέ, αλλά πολλές φορές αυτό συμβαίνει και σε επίπεδο εθνικών εκλογών. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προτείνουμε να ανοίξει δυνατότητα για ψηφοφορία μέσω ίντερνετ ή διαζευτικό ή και ε, μέσω ταχυδρομείου, ταχυδρομική ψηφοφορία για όσους τη στιγμή της ε, ψηφοφορίας δεν βρίσκονται στο χώρο κατοικίας τους, στη χώρα κατοικίας τους. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, το όριο των 16 ετών ε, μου δημιουργεί πρόβλημα. Στο Λουξεμβούργο μόλις τελείωσε μια, ένα ε, δημοψήφισμα στο οποίο καταψηφίστηκε ε, με ποσοστό 80% η δυνατότητα ε, να ψηφίζουν οι νέοι στην ηλικία των 16. Και οι νέοι ακόμα το απέρριψαν αυτό. Πάντως ήταν νομίζω μία από τις κακές ιδέες που συμπεριλήφθησαν και θα ήθελα να μείνει εκτός. Ξέρω γιατί βιαζόμαστε και πιστεύω πως έχετε δίκιο γιατί αν πραγματικά θέλετε να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα στο Συμβούλιο θα πρέπει να γίνει κατά την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να σας συγχαρώ και εσάς και τον Γιώ Λάινεν για όλη αυτή την εξαιρετική εργασία που κάνετε στα πλαίσια της πρότασης αυτής. Αν δούμε λίγο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς εξελίχθηκαν οι εκλογές ε, του 2004. Ξέρετε ότι στην ε, Κροατία είχαμε δύο εκλογές ε, σε δύο-τρεις μήνες μόνο, πάρα πολύ κοντά δηλαδή. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε κι εμείς κάποια πράγματα. Θέλουμε όντως να εμπλακούν περισσότεροι πολίτες. με μια συμμετοχή της τάξης όμως του 42-43% όντως θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και αυτό ισχύει ιδίω για τις νέες χώρες που έχουν ε, μικρότερη εμπειρία και αν θέλετε λιγότερα πολιτικά αντανακλαστικά για κάποιες ευρωπαϊκές εκλογές και ευρωπαϊκά ζητήματα που δείχνουν πολύ συχνά ιδιαίτερα απόμακρα. Νομίζω λοιπόν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να φέρει πιο κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες θα πρέπει να υποστηριχθεί. Και υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο ως προς το οποίο οι εθνικές μας νομοθεσίες αποκλείουν αρκετά. Η χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας, κάτι το οποίο δεν θίξατε καθόλου. Το ανώτατο όριο που προβλέπεται στην εθνική μας νομοθεσία για μία εκλογική εκστρατεία 50 ημερών για ένα σύστημα αναλογικής είναι 200.000 ευρώ για το σύνολο του εκλογικού καταλόγου, για το σύνολο της λίστας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν κατάφερε κανείς από τους υποψηφίου να κάνει τηλεοπτική καμπάνια για παράδειγμα. Και ένα 75% τελικά των ψηφοφόρων μείνανε στο σπίτι τους γιατί ακριβώς δεν είχε προβληθεί αρκετά η εκλογική αυτή δικασία. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε και μια κάποια εναρμόνιση όσον αφορά την ίδια τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατιών. Εγώ όπως σας είπα χρειάστηκα δύο φορές μέσα στο ίδιο έτος να ασχοληθώ με προεκλογικές καμπάνιες και νομίζω ότι η προβολή της ίδιας της καμπάνιας, η προβολή των ίδιων των εκλογών είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε επίσης και τους υποψηφίους εκείνους οι οποίοι θα θέλουν να ε, υποψήφοι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο η εκτελεστική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν πιο δημοκρατικά υπόλογη, θα ήταν πιο υπεύθυνη. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να γίνει υποχρεωτικά, αλλά θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε κάτι τέτοιο με την έκθεσή μας. Όσον αφορά την ελάχιστη ηλικία των 16 ετών, κοιτάξτε, το ζήτημα είναι αρκετά λεπτό και ευαίσθητο. Υπάρχουν πολλές εθνικές νομοθεσίες όπου όσοι είναι κάτω των 18 δεν μπορούν να συμμετέχουν σε καμία απολύτως εκλογική διαδικασία. Το να ενθαρρύνουμε αυτή τη στιγμή σε τέτοιες χώρες νέους κάτω των 18 να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές εκλογές ενδεχομένως να είναι κάπως παρακινδυνευμένο, καθότι οι νέοι αυτοί μπορεί να μην γνωρίσουν απολύτως τίποτα όσον αφορά την ίδια την εκλογική διαδικασία αλλά και την ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι λίγο περίεργο θεωρώ να μην μπορεί κανείς να ψηφίσει για τις εθνικές εκλογές ή για τις δημοτικές εκλογές, αλλά από την άλλη να μπορεί να ψηφίζει για τον υποψήφιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή για την εκλογή Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω λοιπόν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά αυτή την πρόταση. Κάτι το οποίο συζητήσαμε σε μια προπαρασκευαστική συνεδρίαση είναι η ίδια η φύση της εντολής ενός Ευρωβουλευτή όντως δεν θα μπορεί να λαμβάνει εκτελεστικές αρμοδιότητες και στη συνέχεια να μπορεί να επιστρέψει στην ε, θέση που έχει εδώ πέρα ως Ευρωβουλευτής. Νομίζω ότι ιδίω όταν χρησιμοποιείται το σύστημα το προτιμησιακό είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ποιε είναι οι δυνατότητε οι οποίε υπάρχουν για να ευρωβουλευτεί και αν μπορεί τελικά κάποιο ο οποίο έχει συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση ή στην εκτελεστική εξουσία να επιστρέφει στη συνέχεια και να λαμβάνει μια θέση, μια έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το δούμε ιδίω στα πλαίσια του προτιμησιακού εκλογικού συστήματος. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όντως να επεκτείνουμε και την προθεσμία έγκρισης για τον Σεπτέμβριο και είναι σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε ένα ισορροπημένο σύστημα εκλογικό ιδίως όσον αφορά αυτή την μειούμενη εκπροσώπηση ιδίως για το σύστημα αυτό το οποίο συζητάμε εδώ πέρα. μετά όλα στις ευχαριστίες Θέλω και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους συζητητές και να χαιρετήσω τις προτάσεις. Ακούστηκε κάπου ο χαρακτηρισμός για την Επιτροπή μας ε, ότι είμαστε η Επιτροπή των Ανοιροπόλων. Νομίζω ότι μπορούμε να θέλουμε να κάνουμε αλλαγές προς το καλύτερο με τρόπο συνετό και επαφή με την πραγματικότητα για να είναι και υλοποιήσιμες αυτές οι προτάσεις πολιτικά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι δυνατόν αυτό. Πού βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε να κάνουμε με μία ε, ελάχιστη εναρμόνιση των εκλογικών διατάξεων γιατί ναι βεβαίως είναι διαφορετικές οι διαδικασίες αλλά κοινή η διεξαγωγή των εκλογών και μετά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την ε, συμμετοχή του πολίτη και την επιλογή του. Πώς λοιπόν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό με την ε, συμμετοχή με ελάχιστους κανόνες, με κριτήρια προσεκτικά, συνετά, με μία επιλογή άνω των 26 υποψηφίων, που σημαίνει ταυτόχρονα και να μην ξεπερνούμε όρια και να μην προξενούμε στρεβλώσεις. Για την άσκηση λοιπόν των πολιτικών δικαιωμάτων είναι απαραίτητο ο Ευρωπαίος πολίτης να μπορεί να ψηφίσει και όταν βρίσκεται σε τρίτη χώρα ηλεκτρονικά, με επιστολική ψήφο όλα αυτά είναι σημαντικά αλλά η πιο σημαντική αλλαγή από τις προτινόμενες είναι αυτή η οποία επιτρέπει να καταστεί πιο ορατή η υπαγωγή σε πολιτικά κόμματα στις ευρωεκλογές γιατί αυτό θα βλέπει στο ψηφοδέλτιο ο πολίτης. Αυτό θα φέρει την πιο ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τις ευρωεκλογέ. Εν προκειμένου λοιπόν και σε σχέση με την ορατότητα των πολιτικών, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που θα εμφανίζονται και στο εκλογικό υλικό αλλά και στο ψηφοδέλτιο πρέπει πέραν αυτής της ορατότητας που θα έχουμε στο έντυπο υλικό το σχετικό με τις εκλογές η ορατότητα να είναι ε, δεδομένη και στην παρουσίαση των υποψηφίων και των κομμάτων τους στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και τα λοιπά μέσα που θα επιτρέψει έτσι στον πολίτη να αντιληφθεί και τη σημασία των ε, εκλογών. και να αντιληφθεί ότι με τη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ εξακολουθεί να ασκεί το δημοκρατικό του πολιτικό δικαίωμα αλλά μέσα σε ε, ευρωπαϊκές διαστάσεις. Ο κύριος Στάνεμανς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω Ολλανδικά. Η πολιτική μου ομάδα γνωρίζει ότι βρισκόμαστε μία μέρα μετά το δημόσιο διάλογο για την ε, ταυτότητα την ευρωπαϊκή. Είμαστε μετά μια ιστορική μέρα όπου βλέπουμε πως γέρνει η πλάστικα πλέον προς τις εθνικές ταυτότητες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί Εξετάζω τις προτάσεις σας. Δεν είναι ακραίες ευτυχώς. Θα ήταν λάθος αυτό. Δεν είναι και πολύ άριθμες. Ε, κάποιες μπορεί να φαίνονται αθώες αλλά δεν είναι όλες. Το κατόφλι παραδείγματι, το εκλογικό όριο δηλαδή για την είσοδο στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο ή ο λόγος για εθνική εκλογική περιφέρεια. Εμείς στο Βέλγιο θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Επαραδείγματι θα έχουμε μια γαλλόφωνη, μια φλαμανδική εκλογική περιφέρεια ανάλογη με την κατανομή την εθνική. Δεν θα πρέπει να γίνει σεβαστή και η εθνική ταυτότητα. Μπορεί να μιλάτε για εναρμόνιση, αλλά νομίζω ότι παρεμβαίνεται στην εθνική ταυτότητα και σε ζητήματα εθνικής αρμοδιότητας. Εγώ δεν υποστήριζω την ιδέα για ευρωπαϊκές ομάδες ή κόμματα, όσο και αν θεωρείτε εσείς ότι έτσι προάγεται τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Αντιθέτως, νομίζω ότι μπορεί να φέρει το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Θέλετε να προβάλλετε λύσεις με λογότυπο και όνομα Ευρωπαϊκού Κόμματος πάνω στα έντυπα. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε επί της ουσίας τι κάνει και τι δεν κάνει η Ευρώπη. Ποιο είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να είναι πιο συν ομοσπονδιακή, πιο περιορισμένη και όχι τόσο διευρυμένη όπως εσείς ζητάτε επιμόνως. Ζητώντας μάλιστα τώρα ε, ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο. Και αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε να ολοκληρώσω. Για τη συμμετοχή. Κοιτάξτε, το δημοψήφισμα αποτελεί το άκρον άοτον της δημοκρατικής συμμετοχής για τον πολίτη. Το χτεσινό δημοψήφισμα λοιπόν Βλέπουμε να το απορρίπτει ο ίδιος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος συμμετείχε στην εκστρατεία υπέρ του ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή των Σταγματικών ε, Υποθέσεων έχει, θα έπρεπε, θα όφυλαν να ε, δείξουν πολύ μεγάλη σύνεση και περισυλλογή και ταυτόχρονα να περιμένουν για να εκδηλώσουν, να αντιδράσουν στο τελικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Η Μάιτε. Μιλάμε για την εθνική ταυτότητα. Πιστεύω πως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο θέμα αυτό. Και μία από τις μεγάλες απειλές για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι η, κατα η έννοια της εθνικής ταυτότητας που θα ερμηνεύεται με πάρα πολύ περιοριστικό και στενό τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε που θα πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων. όλων. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά εδώ και κάποιοι πιστεύουμε πως θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Τα κράτη, κάποιος μας πριν από 60 χρόνια, είναι υπερβολικά μικρά για να μπορούν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των επόμενων γενεών. Και υπάρχουν θέματα ουσιαστικά που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε, που βέβαια θα αλλάξουν τα ήθη και τα έθιμα. Έχουμε κάποια σύμβολα όλοι μέσα μας, τα οποία ίσως χρειαστεί να μετατρέψουμε Εμένα δεν μου αρέσουν οι εθνικισμοί και αν δεν ξεπεράσουμε τους εθνικισμούς δεν θα ξεπεράσουμε τα διέξοδά μας ανεξάρτητα αν προερχόμαστε από ένα μικρό ή ένα μεγάλο ε, έθνος. Οι μεταρρυθμίσεις που μπορούμε να προτείνουμε θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι η προσβασιμότητα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα υπάρχουν τεχνικές λύσεις και έτσι μπορεί κάποιες ε, κοινωνικές ομάδες να έχουν μεγαλύτερο ή διευρυμένο δικαίωμα συμμετοχής. Για την ηλικία των νέων και πότε θα μπορούν πια να ψηφίσουν, εδώ υπάρχει μια εσωτερική αντίφαση. Θα ήθελα καταρχήν η εκπρόσωπο τη ομάδα μου, η Σιλβή, να ευχαριστήσει του συζητητέ και να πει πω γενικά θεωρούμε πω η κατεύθυνση που ακολουθείτε είναι ε, σωστή, αλλά πρέπει να σα πω πω προσωπικά τα 16 χρόνια μου φαίνονται λίγα. Θα μπορούσε βέβαια αυτό να βοηθήσει να δημιουργηθεί μια τάση οι νέοι στα 14-15 να προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνει η ευρωπαϊκή πολιτική, πώς είναι ο κόσμος που οικοδομούμε, αυτό ναι θα συνέβαινε, αλλά δεν ξέρω αν στα 16 είναι η κατάλληλη ηλικία για να μπει κανεί ε, σε μια ψηφοφορία με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Να το διαπραγματευτούμε όμως, να δούμε τις λεπτομέρειες. Πάντως αποτελεί μια καλή αρχή, μια θετηρία έτσι ώστε να έχουμε ένα οικοδόμημα ε, ευρωπαϊκό που θα αποτελέσει λύση για τα προβλήματα και όχι εμπόδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για όσες προσπάθειες κάνατε. Ευχαριστώ ε, Μάιτε. Ο Μαξ Άντερσον είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω με ευχαριστίες προς τους εισηγητές για τα όσα έκαναν. Έχω τρία σχόλια που θα ήθελα να κάνω. Εγώ παρακολουθώ τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων γιατί είμαι ο παδός της πολιτικής. Μην εκπλήσεστε λοιπόν που παρακολούθησα τις ειδήσει από το ελληνικό δημοψήφισμα εχθές υπάρχει κάποια παρατήρηση που θα κάνω που συνδέεται με τα όσα έχουμε στην ε, δική μας ε, έκθεση. Ήτανε, δεν είχαμε exit poll χθες, είχαμε δημοσκοπήσεις που ελήφθησαν χθες και τα τέσσερα από αυτά τα exit poll μίλησαν για πολύ μικρή διαφορά. Τέσσερις τέτοιες δημοσκοπήσεις είχαμε για κάποια ε, βραδιά η οποία θα είναι πραγματικά έντονο συγκινήσεων και τελικά όταν είδαμε τα αποτελέσματα είδαμε πως τελικά δεν είχαν πετύχει. Δηλαδή ήταν μάλλον σαν μια υποδρομία με ξεκάθαρο ηγέτη της κούρσας από την αρχή. του 61 ήταν πολύ μεγάλη διαφορά με το 39 ε, και πρέπει να σας πω πως έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ε, στο ότι μετρήθηκαν σωστά οι ψήφοι στο ελληνικό δημοψήφισμα αλλά φανταστείτε, φανταστείτε να ήταν η ηλεκτρονική η ψηφοφορία στην περίπτωση αυτή τι θα έλεγαν οι αιτημένοι όποιος και να έχει αιτηθεί δεν θα είχαν εκτοξευθεί κατηγορίες για το γεγονός πως έγινε πως ήταν τεράστια διαφορά μεταξύ exit poll και της καταμέτρησης και πως χρειάζεται ε, έρευνα, μήπως υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Και αυτό θα ήταν φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές μεταξύ ε, δημοσκοπήσεων, exit poll και αποτελεσμάτων. Αλλά οι πόνοιες που δημιουργούνται όποτε υπάρχουν τέτοιες μεγάλες διαφορές με τα πραγματικά αποτελέσματα θα υποσκάψει την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία στις χώρες που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί στο σημείο αυτό, γιατί θα υποσκάψει τη δημοκρατία, γιατί ο κόσμος δεν θα εμπιστεύεται τους υπολογιστές να έχουν κάνει σωστή καταμέτρηση. I'm Έχω και ένα δεύτερο που θα ήθελα να, σας, ε, να μοιραστώ μαζί σας. Γιατί 26, γιατί 26 ευρωβουλευτές, γιατί τέτοιου είδους κατόφλοι. Μπορώ να φανταστώ την εύκολη απάντηση που υπάρχει, αλλά ε, απλώς κάνω την ερώτηση. Και θα ήθελα να ρωτήσω και το εξή. Η πρόταση που έγινε για τα λογότυπα και για τα ονόματα των ευρωπαϊκών ε, κομμάτων και το κατά πόσο θα πρέπει να βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο. Δεν νομίζω ότι η πολιτική ομάδα είναι πιο σημαντική από το Ευρωπαϊκό Κόμμα και για το κατά πόσο μπορεί να φανταστεί μετά ο Ευρωβουλευτής πώς θα ψηφίσει, αλλά νομίζω πως υπάρχει πρόβλημα εδώ. It's going to confuse people on how they are going to vote. Νομίζω ότι στη Σουηδία, για παράδειγμα, εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα με ενστάσεις πολιτών που πήραν το λάθος ψηφοδέλτιο. Γιατί το όνομα κάποιου κόμματος ήταν παρόμοιο με κάποιου άλλου. Και τα ψηφοδέλτια αυτά, ξέρετε, των μικρών κομμάτων για να προκαλέσουν σύγχυση στους ψηφοφόρους ε, προσωμιάζουν στα ψηφοδέλτια των μεγαλύτερων κομμάτων. Καταλαβαίνετε πως αυτό δεν διευκολύνει τον πολίτη να ψηφίσει. Και υπάρχει ένα θέμα αρχής εδώ. Έχουμε εδώ το λογότυπο του Εθνικού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κόμματος στο ψηφοδέλτιο. Θα δημιουργήσουμε σύγχυση για το κατά πόσο ψηφίζουν το εθνικό πρόγραμμα ή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του κόμματος. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κυρία Κωνστανσου, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω, όπως και οι προηγούμενοι, εσάς και τον Γιολάινεν για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση εκθέσεως. Πολύ σύντομα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο, μου επιτρέπετε. Μια ναι, και έχουν ακούσει τόσα πολλά ενδιαφέροντα και ποικίλα από τους προλαλήσαντες. Το σημείο στο οποίο γίνεται λόγος για την ε, εξισορρόπηση μεταξύ των φίλων στην εκπροσώπηση, στην παράγραφο 12. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους της Επιτροπής των Σταγματικών Υποθέσεων Ίσως να γνωρίζετε βέβαια ότι υπάρχει μια πρόταση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ε, μια οριζόντια πρόταση που σημαίνει την εισαγωγή με τροπολογίες ε, προτάσεων σε διάφορα νομοθετήματα από την Επιτροπή των Γυναικών σε συνεργασία και με την Επιτροπή των Σταγματικών Υποθέσεων. Εγώ εκ μέρους Επιτροπής των Γυναικών έχω επιφορτιστεί με την υποβολή της σχετικής προτάσεως στην Επιτροπή των σχετικών προτάσεων στην Επιτροπή των Γυναικών για την ε, ενσωμάτωση της έστασης του φύλου στα νομοθετήματα και αυτή τη στιγμή ασχολούμαι εις βάθος με το θέμα αυτό χωρίς να θέλω λοιπόν να προδικάσω τις όποιες εξελίξεις σε σχέση με μια ενδεχομένη συμφωνία με τους αδέλφους, θα υπάρξουν τροπολογίες για τη διάσταση του φύλου, σχετικές με τη διάσταση του φύλου από την Επιτροπή των Γυναικών. Χωρίς, όπως είπα, να μπορούμε να προδικάσουμε την κατεύθυνση προς την οποία θα βαίνουν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα είναι πάντως αρκετά μαχητικές και συγκεκριμένες σε σχέση με τις ε, ε, προτάσεις ή καλύτερα τις αιτιολογικές σκέψεις του σημείου 12. Και θα τα δούμε βέβαια πάλι και στην Επιτροπή των Γυναικών και εδώ στην Συνταγματική Επιτροπή όπου πιστεύω ότι θα περάσουν αυτές οι τροπολογίες της Επιτροπής των Γυναικών, φιλόδοξες ελπίζω. Σε λίγες μέρες θα έχω να σας δώσω πιο πολλά στοιχεία, ήθελα να σας ενημερώσω πλέον. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Πρέντα να σας συγχαρώ και εσάς και τον Γιολάινεν για την πολύ ποιοτική αυτή έκθεση. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι στην έκθεση αυτή κάνετε προτάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στα δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Το πρώτο είναι ότι δεν έχουμε ότι δεν έχουμε μία ομοιόμορφη ευρωπαϊκή εκλογή αλλά 28 διαφορετικές ε, ευρωπαϊκές εκλογές και πολλές φορές ερμηνεύονται οι εκλογές αυτές ως μια δοκιμή για την ε, κυβέρνηση σε κάθε χώρα ή πολλές φορές αποτελούν ευκαιρία για διάφορους, ε, διάφορες ακραίες πολιτικές δυνάμεις να στραφούν κατά της ίδιας της Ευρώπης και είναι γνωστά τα αποτελέσματα σε κάθε κράτος μέλος βέβαια και γνωρίζουμε τι γίνεται μετά από τις εκλογές αυτές σε πολλά κρατημέλη και πώς τελικά κερδίζουν έδαφος πολλές φορές οι λαϊκίστικες πολιτικές ομάδες. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της συμμετοχής που παρουσιάζει μείωση στις περισσότερες χώρες μολονότι βέβαια στις τελευταίες εκλογές είχαμε την ίδια συμμετοχή με αυτή που είχαμε πριν από πέντε χρόνια. Συμφωνώ λοιπόν με τις προτάσεις που κάνετε, βρίσκονται σωστή κατεύθυνση και έχουν ως απότερο στόχο να έχουμε μία προσέγγιση των 28 διαφορετικών συστημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και από την άλλη προσπαθείτε να ενθαρρύνετε την μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και έχετε υποβάλει εδώ πέρα πολύ καλές ιδέες όπως για παράδειγμα οι 12 αυτές εβδομάδες προθεσμία όσον αφορά τους εκλογικούς καταλόγους, προθεσμία 12 εβδομάδων επίσης όσον αφορά τους επικεφαλείς τη κάθε λίστα, οι οποίοι θα είναι και υποψήφοι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, θέλετε να εμφανίζεται περισσότερο ο λογότυπος των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων σε κάθε ψηφοδέλτιο και λέτε επίση ότι Θέλετε να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιώντας και άλλες μεθόδους όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο. Όλες λοιπόν αυτές οι προτάσεις θεωρώ ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, ότι όντω έχουν ως στόχο να επιλύσουν τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Ας μην έχουμε όμως την ψευδέστηση ότι η προσέγγιση αυτή μεταξύ των 28 διαφορετικών εκλογικών εθνικών συστημάτων θα επιλύσει το πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι αρχικά είχαμε υποβάλει και μια πολύ φιλόδοξη ιδέα το να έχουμε και διασυνοριακές λίστες. Αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι θεωρώ, καθότι δεν γίνεται τέτοια αναφορά στο κείμενο. Αν όμως είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι, ελοχεύει ο κίνδυνος οι ε, πιο ρισπαστικές δυνάμεις να κερδίσουν πάλι έδαφος. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ότι ε, Έχουμε έναν πολιτικό, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής αυτή τη στιγμή και βέβαια προτού γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, ε, είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός μέσω του νέου αυτού συστήματος των Candidate, των ε, υποψηφίων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει τώρα και μετά το ελληνικό δημοψήφισμα, πάντως σε κάθε περίπτωση Είμαι υπέρ όλων αυτών των προτάσεων που θεωρώ ότι ανταποκρίνονται στα δύο αυτά βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και προφανώς θα στηρίξουμε και οποιαδήποτε άλλη τροπολογία κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. σύγκληση των 28 διαφορετικών εθνικών συστημάτων εκλογής που έχουμε αυτή τη στιγμή και παράλληλα ενθάρρυνση της συμμετοχής στις εκλογές, ενθάρρυνση των Ευρωπαίων πολιτών να πάνε να ψηφίσουν. Αν δούμε για παράδειγμα τους Εστονούς που θεωρώ ότι έχουν το καλύτερο σύστημα παγκοσμίως όσον αφορά την ηλεκτρονική ψήφο. Αν υιοθετούσαμε ένα τέτοιο σύστημα θα βρισκόμασταν και εμείς σε πολύ καλύτερη θέση. Αυτό το σύστημα ε, υιοθέτησαν οι Εστονοί και έχουν καταφέρει να επιταχύνουν το σύστημα και να βρουν και μία λύση στο ζήτημα αυτό της ταυτοποίησης των ε, ε, συμμετεχόντων, του εκλογικού σώματος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους ηγητές για την έκθεση. Ασχολείται με πολλά σημαντικά θέματα, θα καταθέσουμε τροπολογίες. Δεν επισέρχομαι τώρα στις λεπτομέρειες, για να είμαι σύντομος. Πρέπει όμως να πω ότι δεν φοβόμαστε καθόλου τις σοβαρές, τις σημαντικές αλλαγές. Δεν είμαστε κατά αυτή τη ενία συντηρητικοί. Δεν φοβόμαστε τις αλλαγές. Αν θέλουμε να φτιάξουμε, να κατασκευάσουμε μια καλύτερη Ευρώπη πρέπει να δείξουμε θάρρος. Πρέπει να προχωρήσουμε με ενθουσιασμό. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που πρότειναν παρατεταμένη προθεσμία για τις τροπολογίες αυτό με το οποίο διαφωνώ είναι με μια παρατήρηση του Ραμών που έκανε δύο σχόλια κατά τη γνώμη μου εσφαλμένα και γι' αυτό το δηλώνω εδώ. Δεν είναι αλήθεια πως αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η κυριαρχία ανήκει στην ίδια την Ευρώπη γιατί πολλές φορές το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν αυτού του είδους την κυριαρχία που έχουμε σε εθνικό επίπεδο και νομίζω ότι η συζήτηση που κάνουμε εδώ είναι ακριβώς η απόδειξη αυτού γιατί δεν υπάρχει ακόμα η ομόσπονδη Ευρώπη και επίσης κανένα κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε η Ελλάδα μπορεί να κάνει κάτι ε, από μόνη του οι πολίτες απλώς εκφράζουν την άποψή τους. Και αυτό κατόπιν συμφωνείτε, συζητείτε με τις απόψεις των υπολείπων. Άρα λοιπόν δεν είναι κίνδυνος αυτό το οποίο εσύ περιέγραψες με το να γίνονται δημοψηφίσματα στην Ευρώπη και ξέρει πολύ καλά που αναφέρομαι μου φαίνεται απολύτως δημοκρατικό ο κόσμος να εκφράζει τη γνώμη του και αυτή να γίνεται ακουστή. Ευχαριστώ πολύ, λέω Παύλο. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος να δηλώσω πως είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τις προσπάθειες που έκαναν οι δύο εισηγητές Στο τελευταίο έγγραφο νομίζω με την τελευταία εκδοχή του έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Ίσως το πρώτο να ήταν πρώτη εκδοχή να ήταν πιο ενθουσιώδης αλλά λιγότερο ρεαλιστική και θα ήταν δύσκολο να εφαρμόστεί στην ε, πράξη. Ακόμα και να συμφωνούσαμε πολλά από τα σημεία που είχε τότε, προτιμώ να έχουμε μια πράξη η οποία θα εφαρμοστεί παρά με το να έχουμε μόνο κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες απλώς χρησιμοποιούνται προς προβληματισμό. Να τονίσω μόνο ή μάλλον να σταθώ σε δύο σημεία όπου διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα το όριο ηλικία των 16 ετών. Νομίζω πως πως δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Θα δημιουργούσε λοιπόν προβλήματα αυτό το συγκεκριμένο όριο, όχι πως δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Και δεύτερον, κατανοώ απόλυτα τη σημασία που έχει ιδιαίτερα για κάποια κράτη να μπορούν να συμπεριλαμβάνουν ένα κατόφλι. Δεν θα εθέσπιζα αυτή την υποχρέωση αλλά θα το άφηνα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν σε εθνικό επίπεδο τι θα ισχύσει. Κάποια κράτη-μέλη έχουν κάποια πλειοψηφικά συστήματα, άλλα κράτη ακολουθούν το αναλογικό. Ας το αφήσουμε λοιπόν στα κράτη-μέλη το θέμα αυτό. Έχω δύο αμφιβολίες που σχετίζονται με ένα θέμα το οποίο δεν είμαι σίγουρος πως κατανόησα καλά. Το, η πρώτη διευκρίνηση έχει να κάνει με το θέμα στη σελίδα 7, το σημείο 10. Να δούμε τη συμφωνία πλαίσιο και να την αναθεωρήσουμε για να δούμε ποια θα είναι η θέση των επιτρόπων. Τι σημαίνει αυτό. Θέλουμε οι επίτροποι να ασκούν καθήκοντα μέχρι και τη στιγμή της εκλογής ή ζητάμε να αναλαμβάνουν έναν άλλο ρόλο ο, κατά τη διάρκεια της εκλογής διαδικασίας. Και υπάρχει και ακόμα κάτι που δεν ξέρω αν είναι λάθος εδώ ή αν εγώ σφάλω. Στην τροπολογία 11 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέμε που αποφασίζει ποια θα είναι η εκλογική περίοδος και ορίζει μία περίοδο 12 εβδομάδων. Νομίζω πως είναι ένα έτος. Οπότε εδώ έχουμε μία μεγάλη μείωση. Εδώ έχουμε ένα μήνα. Με συγχωρείτε, εδώ έχουμε αυτές τις... Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ένας μήνας. Είναι ένα έτος. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε εκλογική περίοδο 12 εβδομάδων, τι κάνουμε. Ουσιαστικά μειώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις προθεσμίες. Εν δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει. Έχω την εντύπωση πως όταν το Συμβούλιο ορίζει ποιες θα είναι οι, οι εκλογικές ε, ημερομηνίες το κάνουν ε, ένα χρόνο νωρίτερα και όχι ένα μήνα νωρίτερα. Άρα λοιπόν νομίζω στην τροπολογία 11 χρειάζεται να κάνουμε μια μικρή διόρθωση ή διευκρίνηση. Thank you. I, uh, Yo, you will... Ευχαριστώ Γιώ, θες να δώσεις απαντήσεις. Εσύ πρώτα γιατί πρέπει να φύγεις για την άλλη μέλη. Ναι, καταρχά ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσει. Εκφράστηκαν με μεγάλη ειλικρίνεια οι θέσεις. Η συζήτηση αφορά βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμα και όταν δεν θα είμαστε εμεί εδώ θα υπάρχουν ευρωεκλογέ, επόμενε, μεθεπόμενε. Και εμεί θέλουμε να βελτιώσουμε το σύστημα και να δώσουμε στου πολίτε ένα καλύτερο, πιο διαφανέ σύστημα και την ευκαιρία και τη βούληση να, να συμμετέχουν σε αυτά τι εκλογικέ αναμετρήσει. Θα απαντήσω λοιπόν ε, ως προς ε, τα δύο στάδια στα οποία αναφέρθηκα για τι μεταρρυθμίσει, ότι τα επιλέξαμε ακριβώς για να επιτύχουμε το στόχο μας. Η Περβόνς Μπερές με ρώτησε, μα αυτό δεν ήταν ένα πάγιο ζήτημα που πάντα προέκυπτε επιτάπητος κάθε φορά που ερχόντουσαν ευρωεκλογέ. Μα ακριβώς αυτό είναι και γι' αυτό διαλέξαμε σε δύο στάδια τη διαδικασία για να ξεκινήσουμε με την δυνατότητα υλοποίηση μιας νομοθετικής πράξης. Άλλωστε και με την έκθεση Φερχόφστατ πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται να κατατεθούν θαραλέες προτάσεις για αναθεώρηση των συνθήκων. Ασχέτως όμως ή αποκομμένες από την νομοθετική πράξη θα έχουμε αυτές τις συστάσεις, τα 13 αυτά σημεία, εν μέρη συστάσεις, που όμως και πάντως δεν ανήκουν, δεν εντάσσονται στο κείμενο της νομοθετικής πράξης. και αναλόγως μπορούν να την Η κυρία Λογκρίπ, ε, ο κύριος Λογκρίπ μας λέει ότι πρέπει να περιμένουμε, όχι η κυρία Λογκρίπ μας λέει ότι πρέπει να περιμένουμε τι θα προκύψει από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών σε σχέση με τις ε, τροποποιήσεις, με τις τροπολογίες που θα καταθέσει την ΑΦΚΟ για την ε, ενσωμάτωση διάσταση του φύλου. Την ξεχνάμε ότι πρέπει όμως το Συμβούλιο και να ψηφίσει με ομοφωνία και αυτό σημαίνει να ψηφίσουν όλα τα κράτη-μέλη κατά τρόπον ώστε να περάσει το κείμενο χωρίς να επιβαρυνθεί με τροποποίησεις τέτοιες που θα εξουδετερώσουν τελείως, θα το κενώσουν ε, ενδιαφέροντος και νοήματος. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω για τον κύριο Σέμφλιν όταν μιλούσε για Spitzenkandidaten εννοούσε άραγε ότι οι 12 εβδομάδες δεν αρκούν και ότι χρειάζεται για τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου να προβλεφθεί μια μακρύ, μακροίτερη ε, χρονική περίοδος για να μπορέσει να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία σε όλα τα κράτη. Αν κατάλαβα καλά, πάντως μπορούν να κατευθούν τροπολογίες η δυνατότητα συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία για κάποιον που ζει σε κράτο εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σκεφτώ, α πούμε, τα νησιά Φίτζι που επισκεφθήκαμε ορισμένοι εξημών ή το Μπαγκλαντέ. Φαντάζομαι ότι όλα τα προξενικά ε, καταστήματα έχουν αυτή τη στιγμή εξοπλισμό ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύνδεση στο, διαδίκτυο. Άρα φαντάζομαι ότι εκμηδενίζονται οι αποστάσεις και μπορούν ταχύτητα να διαβιβαστούν τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει πια χιλιομετρική απόσταση. Από την άλλη πλευρά, 9 πρωί έως 9 το βράδυ, 24, 12 ώρες. Αυτό που αναφέρατε εσείς ότι κοιτάξαμε με τι ώρα τελειώνουν οι ε, εκλογές, κλείνουν οι κάλπες, αλλά δεν αναφερθήκαμε στο τι ώρα θα ανοίγουν. Εμείς στη Γερμανία νομίζω ανοίγουμε κάπου στις 8 τις κάλπες. Φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουμε βεβαίω. Και κατά πόσο είναι και χρήσιμο. Κύριος Πλένκοβιτς, αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατείων, θέμα πολύ σημαντικό και αξιόλογο, και το θέμα βέβαια της χρηματοδότησης των κομμάτων, θα θυμάστε ότι είχαμε ένα καταστατικό των ευρωπαϊκών κομμάτων, που παραλίγο να απορριφθεί ακριβώς λόγω του ζητήματος της χρηματοδότησης των κομμάτων γιατί υπάρχουν τέσσερα κράτη στα οποία απαγορεύεται η αδίποτε δωρεά σε πολιτικά κόμματα. Πριν από δέκα χρόνια περίπου παραλίγο να καταρριφθεί, να απορριφθεί αυτή η πρόταση λόγω ακριβώς του θέματος της χρηματοδότησης. Καυτό θέμα, ίσως πρέπει στις συστάσεις να το περιλάβουμε αν θέλουμε οπωσδήποτε να το θίξουμε. Ε, το ασυμβίβαστο και η δυνατότητα επανόδου στις επαγγελματικές δραστηριότητες των ευρωβουλευτών όταν ε, λύγει η θητεία τους. Δεν το έχουμε θίξει καθόλου, το κοιτάξουμε. Μετά, για τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν στο εκλογικό όριο, για τον κύριο Άγγεμανς, για το Βέλγιο δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που διατύπωσε ως υπόθεση. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα το Βέλγιο. Για τον άλλο συνάδελφο είναι 26 ή άλλο. Κάτω των 26 εδρών έχουμε de facto όριο 3%. Στις 26 και άνω των 26 εδρών μπορούμε να έχουμε χαμηλότερο κλικικό όριο 2,5-2,3%. Η Γερμανία έχει 0,5 παραδείγματι. Για εντολή βουλευτική, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε 14 ε, βουλευτικές έδρες με πάρα πολύ μικρό ποσοστό εκλογής, εκλογικό όριο. Το ίδιο έχει και η Ισπανία. Άρα έχουμε ε, μία de facto μη τήρηση του εκλογικού ορίου του 3%. Αλλά όπως είπα αυτό αφορά τις ε, περιπτώσεις όπου έχουμε πάνω από 26 έδρες. Ντανούτα, θα πω τώρα, αυτά είχα να πω. Θα πω ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. 29 Ιουλίου θα ήταν καλό να μείνει η συνεδρία που έχουμε προβλέψει για να αξιοποιήσουμε και την παρουσία της ε, Λουξεμβουριανής Προεδρίας. Είναι καλή ευκαιρία και πρέπει να αξιοποιήσουμε γιατί η επόμενη Προεδρία δεν φαίνεται να φλέγεται τόσο για το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν καλό θα είναι να κοιτάξουμε όσο είναι νωρίς τα θέματα αυτά πριν χαθούν οι ευκαιρίες. Αλλά φαντάζομαι ότι η γραμματεία θα έχει τη δυνατότητα να μας κάνει καλές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ τους ε, συναδέλφους για τη συμμετοχή. Σε ευχαριστούμε Γιώ. Να προσθέσω και εγώ λίγα πράγματα. Ο Ραμόν είπε κάποια στιγμή ότι δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι, μα θα θυμάσαι ότι είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε μέσω ε, εκτελεστικών πράξεων να επιφέρουμε περαιτέρω τροποποίησης. Εμείς όμως επιλέξαμε να τροποποιήσουμε τον ίδιο τον εκλογικό νόμο και μόνο και μόνο αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου. Δεν χρειαζόμαστε μόνο βέβαια αμοφουνία στο Συμβούλιο για να τροποποιηθεί ο νόμος αυτός, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και εξαρτώμενο από την κάθε χώρα προβλέπεται και διαδικασία εθνικής έγκρισης ε, του κειμένου αυτό από τα εθνικά κοινοβούλια. Θελήσαμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας όλη αυτή την πολύπλοκη διαδικασία. Θελήσαμε να συντονιστούμε επίσης με το Συμβούλιο, να δούμε ποια είναι η πρόθεσή τους και βλέπουμε ήδη από τη Λουξεβουργενή Προεδρία ότι όντως θέλουν να δεσμευθούν για να ευοδοθεί η διαδικασία αυτή, γιατί με την επόμενη Προεδρία ενδεχομένω τα πράγματα να είναι λίγο πιο δύσκολα. Και ξέρετε ότι και στην έκθεση του Γκίφερ Φερχόφστατ ε, μέσω τροπολογιών μπορούμε να περάσουμε και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ενδεχομένω να μην καταφέρουμε να περάσουμε την έκθεση αυτή. Είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν κάποιες κέρδιες τροπολογίες όταν ο τίτλος της έκθεσης είναι Ευρωπαϊκός Εκλογικός Νόμος, ενώ νομίζω ότι στην έκθεση Φερχόφστατ υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο περιθώριο τροποποιήσεων. Υπάρχουν επίσης και κάποια ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στον Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο, όπως το ζήτημα της χρηματοδότησης ή το ζήτημα των εν επιτρόπων, ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε εμείς να διευθετήσουμε απευθείας μέσω της έκθεσης αυτής. Πάντως, Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να δούμε και ποιες θα είναι οι τροπολογίε σα. Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε τις τροπολογίες αυτές. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να θέσουμε ως ημερομηνία την 10η Αυγούστου. Ενδεχομένως να μην καταφέρουμε να μεταφράσουμε μέχρι τότε όλες τις τροπολογίε, αλλά αν υποβάλει τροπολογίε μετά τη 10η Αυγούστου, τότε σίγουρα θα τις έχετε μόνο στα αγγλικά. Αν τηρήσουμε την προθεσμία αυτή του Αυγούστου, τότε μπορούμε στις 3 Σεπτεμβρίου να συζητήσουμε τις τροπολογίες αυτές και να έχουν και όλες μεταφραστεί. Συμφωνείτε λοιπόν 10 Αυγούστου προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Μπορείτε όσοι προτιμάσετε πιο γρήγορα τις τροπολογίες να τις στείλετε όπως είπε και ο Λάινεν μέχρι τις 29 Ιουλίου. Διαφορετικά οι υπόλοιποι θα έχετε χρόνο μέχρι τις 10 Αυγούστου. Λοιπόν, η 10η Αυγούστου είναι η προθεσμία σύμφωνα με την οποία μπορείτε να υποβάλλετε σε οποιαδήποτε γλώσσα στην α, μητρική σας γλώσσα της α, και θα τις μεταφράσουμε μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Πάλι θα αναφερθούμε πάντως και στο ζήτημα αυτό για το οποίο εξέφρασες κάποιες αμφιβολίες. Δεν έχω να πω εγώ τίποτα άλλο. Θα υπάρξουν κάποιε νέε τροπολογίε γιο και στο λέω, πράγματα τα οποία σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Πάντω μπορούμε να κλείσουμε τώρα αυτό το σημείο στη μερίσια διάταξη και να περάσουμε στο σημείο 6 όπου θα συζητήσουμε την έκθεση του Γιώργη Σοπφλίν για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Θα μας παρουσιάσεις, αν κατάλαβα καλά, τις τροπολογίες, έτσι δεν είναι? Γιατί περνάμε τώρα στην επόμενη φάση εξέτασης της έκθεσης αυτής, λοιπόν. Ο Γιώργη Σόπφλιν έχει το λόγο. Δεν θα παρουσιάσω όλες τις τροπολογίες γιατί είναι 127 στο σύνολο και η ζωή είναι σύντομη. Αυτό που θα κάνω είναι να σας υπενθυμίσω πως τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το μέσο αυτό είναι πολλά. 51 προσπάθειες ε, έγιναν για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία πολιτών καμία δεν ξεκίνησε στην πράξη. Έχουμε λοιπόν αποτυχία στο 100%. Είναι ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Δεν θεωρώ ότι είναι νεκρό το εργαλείο αυτό. Μπορεί να λειτουργήσει και στην έκθεσή μου προσπάθησα να βρω κάποιους τρόπους έτσι ώστε να σταθεί στα πόδια του. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια μεγάλη αναθεώρηση είτε στα τέλη του της χρονιάς είτε στην αρχή του επόμενου έτους και θα ήθελα οι δικές μας συζητήσεις εδώ και οι δικές σας να επηρεάσουν τη συζήτηση αυτή. Και πρέπει να πω από τις επαφές που είχα πως μάλλον αυτό θα συμβεί. Να πω πως το εργαλείο αυτό, η πρωτοβουλία πολιτών είναι μια καινοτομία μοναδική κατά κάποιο τρόπο και είναι εντυπωσιακό και ο τρόπος που λειτουργεί γιατί το ότι οι πολίτες μπορούν σε έναν ιδανικό κόσμο να κινήσουν μια πρωτοβουλία που οδηγεί τελικά σε νομοθεσία είναι κάτι καινούριο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και θα ήθελα να συμβαίνει 127 τροπολογίες όπως σας είπα σχεδόν όλες είναι χρήσιμες, υποστηρικτικές. Μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη μια-δυο. Γενικά πάντως, ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη αυτής της Επιτροπής και οι υπόλοιποι το αντιμετώπισαν ήταν πολύ θετικό. Σας ευχαριστώ όλους. Και ειδικά όσους υπέβαλαν τροπολογίες. Κάποια προβλήματα σχετίζονται με το ίδιο το εργαλείο είναι το γεγονός πως αυτή τη στιγμή είναι ένα μέσο που δεν είναι φιλικό προς το χρήστη. Θα πρέπει να είναι πιο προσβάσιμο ηλεκτρονικά, δηλαδή για άτομα με αναπορίες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. Ο τρόπος με τον οποίο έχει διαδοθεί το εργαλείο αυτό δεν ήταν πολύ πετυχημένος. Χρειάζεται καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε προς αυτή την κατεύθυνση να τους ενθαρρύνουμε. Με αποτέλεσμα μια καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας με τους πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ένα ζήτημα που προέκυψε και το οποίο στηρίζω απόλυτα είναι πως οι οργανωτές τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα πρέπει να αποφασίζουν σε ποια στιγμή ξεκινά να τρέχει το ρολόι. Δεν θα πρέπει αυτό να γίνεται αυτόματα όπως σήμερα. Και τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Μπορούν οι οργανωτές να συλλέγουν email. Πώς εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων. Η κυβερνοασφάλεια που είναι ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα και έχει συζητηθεί και αλλού η εναρμόνιση στην περίπτωση αυτή των απαιτήσεων για τα δεδομένα σε επίπεδο κρατών μελών είναι ένα θέμα μια και έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα. Δεν είμαι πάντα υπέρ της εναρμόνισης των κανόνων, αλλά εδώ πιστεύω πως αυτό είναι επιθυμητό έτσι ώστε να είναι ίσοι οι κανόνες παιχνιδιού για όλους τους πολίτες. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα δεν μπορούν να υπογράψουν μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Επίσης θα πρέπει να αναλύσουμε την εθνική εμπειρία γιατί ξέρω πως αρκετά κράτη έχουν κάτι αντίστοιχο με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Θα ήταν χρήσιμο να δούμε πώς λειτουργούν αυτά και πρέπει να πω πως οι συζητήσεις που είχαμε τη Λετωνική Προεδρία μίλησα μαζί τους για τις εμπορίες που έχουν είναι μια μικρή χώρα όμως και είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει παρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί δεν χρειάζεται ούτε 7 κράτη-μέλη ούτε ένα εκατομμύριο υπογραφές γιατί αν ε, υπέγραφαν ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη Λετωνία σε ένα συνολικό πληθυσμό 2,5 εκατομμύριο καταλαβαίνετε τι θα συνέβαινε αν αφαιρέσουμε και τους κάτω από τα 16. Το πρόβλημα της χρήσης της μητρικής γλώσσας. Επίσης, αυτή τη στιγμή μπορεί να υποβάλει κανείς μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε μια από τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες γλώσσες που έχουν περιφερειακό ή τοπικό ε, καθεστώς, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα ουαλικά, για παράδειγμα. έτσι ώστε όσοι έχουν αυτή τη γλώσσα ως μητρική να μην βρίσκονται σε μια ανεκτική θέση. Μίλησα με τον Επίτροπο κύριο Τιμέρμαντς και το δέχεται. Επίσης, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πώς συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα πρέπει να συμμετέχουν όμως ε, ιδιαίτερα δραστήρια, θα πρέπει απλώς να παρακολουθούν. Δεν πιστεύω ότι ο ρόλος τους είναι να ηγηθούν τέτοιου είδου πρωτοβουλίες. Έχουμε και άλλες πολλές πρωτο, ε, τροπολογίες που φοβούνται πως μπορούν να χειρογηθούν αυτές οι υπογραφές και το 1 εκατομμύριο αλλά εφόσον είναι στη συνθήκη δεν βλέπω πως θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε δεν νομίζω πως πρόκειται να τροποποιήσουμε τις συνθήκες ε, στο άμεσο μέλλον για το θέμα αυτό Ένα-δύο σχόλια ακόμα. Έχουμε το πειραματικό project για το οποίο μόλις ψηφίσαμε και τη σχετική γραμμή στον προϋπολογισμό, σημαντικό για την προώθηση και κάποιες δυσκολίες στις οποίες θα σταθώ. Πείτε μου τι γίνεται όταν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών διατυπώνεται με στόχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διακόψει κάποιο μέτρο. Μπορούμε να το σκεφτούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και αυτό προέκυψε σε άλλο πλαίσιο, όχι στην πρωτοβουλία. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για το κατά πόσο θα έπρεπε να αλλάζουμε ώρα ε, και να έχουμε θερινή και χειμερινή. Αυτό μπορεί να αποφασιστεί μέσω ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Δεν νομίζω πως είναι παραδεκτό με τους σημερινούς κανόνες. Εγώ για τη θεωρινή ώρα να σας πω πως δεν έχω κάποια άποψη. Ζω και στις τρεις ε, ε, χρονικές ζώνες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά καταλαβαίνετε ότι πάντα υπάρχει πρόβλημα για την υγεία αν κάποιος φεύγει από τη μία ζώνη πέρα από το θερινό ωράριο στο χειμερινό κτλ. I would say we should not be thinking about this, but the, the Petty has voted on this. Ε, νομίζω πως η Επιτροπή Αναφορών έχουν ε, ψηφίσει για το θέμα αυτό. Πιστεύω πάντως πως δεν είναι ρεαλιστικό ε, να προχωρήσουμε κάπου παραπάνω εδώ. Εγώ πάντως πιστεύω πως σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο που να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές ε, διατάξεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά πάντα πιστεύω πως είναι καλή ιδέα γιατί ένα γραφείο το οποίο θα έχει ως μοναδικό καθήκον να βοηθά τους πολίτες με ένα μάλλον περίπλοκο εργαλείο θα βοηθούσε να καλύψει σε κάποιο βαθμό το χάσμα μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ψηφιακή ε, υπηκότητα. Ίσως προηγούμαστε της εποχής μας, θα μπορούσε και αυτό να συζητηθεί. Οι τροπολογίες που έλαβα ε, στο σημείο αυτό είναι μοιρασμένες μεταξύ τους. Κάποιες ομάδες είναι υπέρ, κάποιοι είναι ε, κατά και κάποιες ομάδες είναι μια τελευταία παρατήρηση. Αν γίνει ακρόαση, θα πρέπει να γίνει σε κάποια ουδέτερη επιτροπή. Όχι στην επιτροπή που επηρεάζεται πιο πολύ από την ακρόαση, γιατί τότε υπάρχει ε, πρόβλημα γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις ή συμφέροντα που θα υπερισχύσουν. Οπότε ναι, αν γίνει ακρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να επιλέξουμε μια ουδέτερη επιτροπή ή στην ΑΦΚΟ λοιπόν ή στην ΠΕΤΗ. Ευχαριστώ. Σιλβί. Καφμάν. Yeah. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα προχωρήσαμε. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή. Πολύ καλή η πρόταση του, η πρόταση εκθέσεως και πολύ σαφής η στόχη που περιγράφει. Πρέπει να τροποποιηθεί η πρωτοβουλία των προεπολιτών έτσι ώστε να γίνει και πιο αποδεκτή και πιο εύχρηστη. Έχουμε την εμπειρία αυτή των τριών ετών από την ε, ε, λειτουργία της. Έχουμε δύο-τρεις πρωτοβουλίες πολιτών που κατάφεραν να συλλέξουν το 1 εκατομμύρια των υπογραφών και που όμως δεν συνοδεύτηκαν από το επόμενο βήμα, δηλαδή την πρόταση της Επιτροπής με βάση το αντικείμενο της ε, πρωτοβουλίας πολιτών. Πρέπει λοιπόν να μας αποσχολήσει το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε όλοι μαζί αυτό το εργαλείο. Κοιτάξα τις τροπολογίες και βλέπω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα με περιττέρω συζητήσεις πάνω στα διάφορα θέματα. Θα ήθελα πάντως να αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία τώρα. Γιατί είναι βέβαια μακροσκελής ο κατάλογος των προβλημάτων που έχετε εντοπίσει και εσείς ο ίδιος τοποθετηθήκατε σε αρκετά από αυτά. Ε, θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε το χρόνο να τα συστήσουμε ένα-ένα. Είναι επί παραδείγματι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα το ζήτημα των προθεσμιών για τη συλλογή των υπογραφών, 12 μήνες. Διαφορετικέ ιδέε ακούγονται. Άλλο λέει ότι θα μπορούσε να παραταθεί στου 18 μήνε αυτό το διάστημα. Εγώ θα προτιμούσα ένα διαφορετικό σύστημα ή μοντέλο να είναι διαφορετική, να μην ξεκινάει η προθεσμία με την υποβολή της πρωτοβουλίας αλλά αργότερα. Να μπορούν δηλαδή οι οργανωτές της πρωτοβουλίας να αποφασίσουν ότι έχουν προχωρήσει αρκετά τα οργανωτικά τους ζητήματα και ότι από ένα χρονικό σημείο και μετά αρχίζουν τη συλλογή των υπογραφών και από εκεί και πέρα αρχίζει και τρέχει η προθεσμία για τη συλλογή. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια θετική αλλαγή Βέβαια αυτό σημαίνει και τροποποίηση του κανονισμού, όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα ζητήματα. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να ξανακοιτάξουμε το ζήτημα της μεγαλύτερης δημοσιότητας για την πρωτοβουλία των πολιτών. Σε πολλές εκδηλώσεις, όταν ακούγεται «Α, υπάρχει αυτό το εργαλείο, υπάρχει αυτό το μέσο, η διαδικασία είναι αυτή, χρειάζεται, απαιτείται ένα εκατομμύριο υπογραφές και το καθεξής», Ακούγονται λοιπόν αυτά τα στοιχεία και διαπιστώνω ότι οι ακροατές δεν έχουν ιδέα ότι υπάρχει πρωτοβουλία πολιτών. Ανεξαρτήτως μάλιστα ηλικία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι το ουσιαστικό για να μπορέσει ο πολίτης να πει «Α, ένα λεπτό, εδώ πέρα κάποιος ζητάει τη γνώμη μου και πρέπει και εγώ να τη δώσω, να συμμετάσχω». Σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση και να φροντίσουμε να εξασφαλίσετε υποστήριξη οργανωτές αυτών των πρωτοβουλειών. Το σημείο στο οποίο αναφερθήκατε επί παραδείγματι για τη δυνατότητα παροχής ε, υποστήριξης αρρωγής και συμβουλών για τους οργανωτές αυτών των πρωτοβουλειών είναι μια θετική πρόταση νομίζω. Και επίσης ε, καθόσον μάλλον μεγάλο κομμάτι των πρωτοβουλειών αυτών, το 40% απορρίπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι αναπτύσσονται εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Μια διαδικασία δηλαδή η οποία έχει τις δυσκολίες της και πρέπει να βοηθήσουμε στα νομικά έστω ζητήματα τους πολίτες της Ευρώπης. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο και στα τελευταία ανάλυση ήδη οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν ή όχι. Το άλλο ζήτημα, να γίνουν πιο εύχριστες ή να μειωθούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες η διαγραφή της ε, συλλογής στοιχείων ταυτότητας ε, με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας πάνω απ' όλα που θα απλουστεύσει τις διαδικασίες και που ήταν από ό,τι φαίνεται ένα από τα προβλήματα στη συλλογή των υπογραφών. Μετά ο κύριος Σεμφλίνγκ ε, μας λέει ότι θα καταθέσει τροπολογίες. Εμείς θα έχουμε προτάσεις για την μείωση του ορίου ηλικίας για την συλλογή των υπογραφών. Εγώ πιστεύω και εμείς πιστεύουμε ότι ακριβώς σε ένα τέτοιο σημείο πρέπει να μειώσουμε το όριο ηλικίας και να το πάμε στα 16 έτη. Κάναμε τη συζήτηση μόλις τώρα για το εκλογικό δίκαιο και υπόθηκε ότι το δικαίωμα του εκλέγην από τα 16 ε, χρόνια ηλικίας απερίφθη στο Λουξεμβούργο με δημοψήφισμα. Ναι, έστω αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε την εμπιστοσύνη στους 16 άριδες ότι μπορούν να δώσουν την υπογραφή τους με υπευθυνότητα προς μια κατεύθυνση. Είναι μια ιδέα την οποία θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω λοιπόν. Και τελευταία παρατήρηση. Έχω μια τροπολογία καταθέσει που είναι πολύ σημαντική για μένα κύριε Σούφλιν, θέλω να την κοιτάξετε προσεκτικά. Θέλουμε εκ μέρους μας να, ε, να ε, καταστεί απολύτως σαφές ότι πρέπει να δοθεί ένα τέρμα σε αυτήν την ιστορία του κανονισμού. Υπόθηκε ε, και από εσά κύριε Σοπλήν ότι η Επιτροπή σκοπεύει να καταθέσει πρόταση για αναθεώρηση, για μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση στο τέλος του χρόνου. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να δώσουμε το σχετικό μήνυμα ότι χρειάζεται πλέον αναθεώρηση αυτού του κανονισμού. Πρέπει με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουμε τις θέσεις μας και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια να διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις προς τις κατευθύνσεις που επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας μέχρι τώρα. Προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πρωτοβουλία πολιτών, εύχριστη μια πρωτοβουλία πολιτών που θα ικανοποιεί τον πολίτη. Ευχαριστώ πολύ, Μαϊτέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Σέπφλιν γιατί η δουλειά που κάνετε πραγματικά είναι εξαιρετική, ακολουθεί τη σωστή ε, κατεύθυνση. Θα μοιραστώ με τη συνάδελφο που λείπει τα ζητήματα τα οποία θίξατε. Θεωρώ πως ο φάκελος αυτός είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρος γιατί αυτό που μας παρουσιάζεται είναι πολύ στέρεο και οι τροπολογίες θα το βελτιώσουν ακόμα περισσότερο και θα έχουμε όλη την ευκαιρία να προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες ενδείξεις για το πώς ακριβώς πρέπει να τροποποιήσει τον κανονισμό και την ομοθέσια. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες προσπάθησαν να ξεκινήσουν μια τέτοια της πρωτοβουλία και δεν τα κατάφεραν. Και αυτό δημιουργεί έναν εκνευρισμό που δεν είναι θετικός για τα όσα εμείς προωθούμε. Δηλαδή, το θεματολόγιο των ευρωπαϊκών θεσμών να λαμβάνουν υπόψη τις μεγάλες αυτές προτάσεις που προωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Θεωρούμε επίσης πως θα πρέπει τα εμπόδια τα γραφειοκρατικά να μειωθούν και προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω πως θέλουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, μεγαλύτερη συνειδητοποίηση μέσω κάποιου γραφείου ή οποιοδήποτε μέσο επιλέξετε, έτσι ώστε να έχουμε υπαλλήλους που θα προσφέρουν δεδομένα, που θα επιλύουν τεχνικά ζητήματα, έτσι ώστε από τη στιγμή που θα ξεπερνιόνται τα τεχνικά ζητήματα να μπορεί κανείς να τρέξει την προθεσμία των 12 ε, μηνών χωρίς παρατάσεις ε, γιατί αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Να απλοποιήσουμε μόνο αυτό το οποίο είναι δυνατόν να απλοποιήσουμε και να προωθήσουμε αυτό το οποίο είναι βασικό έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προσπάθεια αυτή των πολιτών όταν το επιθυμούν γιατί ξέρετε πως αυτό θα εμψυχώσει ε, και τη συμμετοχή όλων μας. Εμείς λοιπόν θα σας στηρίξουμε όσο μπορούμε για να τροποποιηθεί η νομοθεσία εδώ, να πλουστευθεί, να είναι πιο υποβοηθητική σε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να εκνευρίζει τους ε, εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Ο κύριος Σέπλιν θα έχει λοιπόν τη στήριξή μας για την προσπάθεια αυτή που σίγουρα θα πάει πάρα πολύ καλά. Ο Χέλμουτ Σόλτς είναι επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστώ τον ε, εισηγητή, πολύ καλή δουλειά του και οι προτάσεις του. Νομίζω ότι προσπαθούν οι συνάδελφοι και με την κατάσταση τροπολογιών να εκφράσουν τις ε, ανάγκες για αναθεώρηση τη νομοθεσία σχετική με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μπορώ να συμφωνήσω λοιπόν πολλά, με πολλά από αυτά που υπόθηκαν σήμερα. Θα επικεντρωθώ όμω σε ορισμένα σημεία μόνο. Νομίζω το σημείο 9 είναι σημαντικό. Τα εμπόδια, τα προβλήματα, προσδιορισμός των ερωτημάτων, όλα αυτά τα οποία καθιστούν τόσο περίπλοκο το εγχείρημα μιας πρωτοβουλίας πολιτών. Και, και δύσκολο επίσης να συλλεγεί υποστήριξη από άλλους πολίτες σε μια δημοκρατική διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να μας αποσχολήσει το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα επόμενο βήμα και νομίζω ότι αυτό καλύπτουν και οι πολυάριθμες τροπολογίες. Πώς θα γίνει πιο πρακτική δηλαδή η υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Για το σημείο 10, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε μια εποχή όπου ε, το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή των πολιτών και της κοινή γνώμης, νομίζω πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώς τα σημεία αυτά. Και δεν είναι και πολλές οι παρατηρήσεις και τροπολογίες που έχουν τεθεί, αλλά πρέπει να τις κοιτάξουμε μέσα από το πρίσμα της επίκαιρης δημόσιας συζήτησης και να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την υποχρέωση για τον οργανωτή της πρωτοβουλίας και την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά τρόπον όμως που να μην είναι τόσο υπερβολικός ώστε να αποτρέπει από την πρόοδο, από την οργάνωση μιας πρωτοβουλίας ε, πολιτών των ενδιαφερομένων Σε αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τον κανονισμό λοιπόν. Επίσης θα ήθελα να συμφωνήσω με το σημείο 13. Υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε μια πρωτοβουλία πολιτών. Θέλουμε λοιπόν να καταστήσουμε δυνατή την πρόοδο για τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες πολιτών αυτές που συνέλεξαν τον επαρκή αριθμό ε, υπογραφών. Όμως πολλές φορές έχουμε συζητήσει και θέματα ε, πρωτοβουλειών οι οποίες, θα, είχαν πάρα πολύ καλή επιτυχία αλλά λόγω του σύντομου των προθεσμιών δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν το 1 εκατομμύριο ψήφους ή παρότι το συνέλεξαν δεν ε, εδόθη συνέχεια. Αυτά όλα πρέπει νομίζω να τα κοιτάξουμε και να βρούμε μια λύση για τροποποίηση των σχετικών σημείων του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σούπλιν και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα θέματα αυτά γιατί είναι αναγκαίο να συζητηθεί το μεγάλο δημοκρατικό αυτό μέσο και εργαλείο που έχει ο πολίτης του να εκφραστεί και πρέπει να το προωθήσουμε, να το αναθεωρήσουμε, να το καταστήσουμε πιο σαφές. Ευχαριστώ κύριε Σκατικάμπρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σέπφλιν για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Πραγματικά εργαστήκατε πολύ καλά. Όλοι θεωρώ ότι εργαστήκαμε πολύ καλά σε σχέση με την έκθεση αυτή και νομίζω ότι θα ευοδοθεί πραγματικά η πρότασή σας αυτή για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού, συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε η συνάδελφος κυρία Κάουφμαν. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, φαντάζομαι Γιώργο ότι αυτοεκτίμησή σε αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευθεί. Λοιπόν, μήπω μπορείτε να, να κλείσετε και σύντομα. Όχι, όχι, δεν έχω απογειωθεί ακόμα. Απλώς να σας πω ότι ε, θέλω να σε ευχαριστήσω και θεωρώ ότι πραγματικά οι παρατηρήσεις αυτές ήταν πολύ επικοδομητικές. Ε, όντως πρέπει να χρησιμοποιείτε καλύτερα το μέσο αυτό, πιο φιλικό προς το χρήστη. Δεν αναφέρθηκα στην ηλικία των 16 ετών, αλλά θα μπορούσα να το δεχθώ και αυτό ως πρόταση. Ξέρετε όμως ότι θα προκαλέσει προβλήματα ενδεχομένω σε κάποιες χώρες, πάντως επί της αρχής δεν θα διαφωνούσα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δούμε τι έχει γίνει στην Αυστρία, διότι στη χώρα αυτή όντως τα πράγματα έχουν κινηθεί καλύτερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Δεν ξέρω τώρα πώς θα τη δράσει βέβαια η Λουξεμβουργιανή Προεδρία και αν θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστριακής. Πάντως εγώ χρειάστηκε να περιμένω να γίνω 21 ετών μέχρι να ψηφίσω. Επομένω, δίστανται πολλέ φορέ οι απόψει για το αν κάποιο είναι όντω έτοιμο όταν είναι 18 ετών. Πάντω, για όλε τι υπόλοιπε παρατηρήσει, σα ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας, για τη συμμετοχή σας, για τις ε, τροποποιήσεις που καταθέσατε και νομίζω ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε και μια συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Στο διάμεσο διάστημα καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την πρόεδρο στις 22 Σεπτεμβρίου. Δεν έχω να κάνω άλλες ανακοινώσει. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 15 Ιουλίου μόνο το πρωί. Τώρα μπορείτε να αποχωρήσετε το συντομότερο δυνατό για να γίνει και η συνεδρίαση των ιστών. Ε, the coordinators have a meeting now, so... Ξεκινήσει σε λίγο συνεδρία των συντονιστών.